Όσον αφορά τις διάφορες αποφάσεις ε, επιτροπών να ξεκινήσουν οργανικές διαπραγματεύσεις βάση του άρθρου 69C παραγραφός 1 που ανακοινώθηκαν στην έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 28 Μαΐου δεν έλαβα αιτήματα ψηφοφορίας ε, από επαρκή αριθμό βουλευτών ή ενός ή παραπάνω πολιτικών ομάδων που είναι ε, με το 10%, επομένως οι επιτροπές μπορούν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει ένα αίτημα από πλευράς του κυρίου Σούλικ για να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας εχθές για την πρόταση αναθεώρησης οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων, δεν καταλάβαμε τι ψηφίσαμε. Γι' αυτό, βάσει του άρθρου 148α, θα ήθελα ε, να προβάλλω μια ένσταση διαδικαστική για τη χθεσινή ψηφοφορία για αυτή την έκθεση. Ο Προεδρεύων έκανε την ψηφοφορία ε, με τρόπο που οδήγησε σε 37 διορθώσεις ε, ψηφοφορίας από τις πολιτικές ομάδες. Αυτό είναι πρωτοφανές παρά το γεγονός ότι είναι αμφιλεγόμενη η πρόταση και παρά το γεγονός ότι κάποιος συνάδελφος από το ΕΛΚ μετά την ψηφοφορία ε, το ζήτησε, ο Πρόεδρος δεν άλλαξε θέση και δεν επανέλαβε την ψηφοφορία. Παρακαλώ να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφοι, όμω πρέπει να σα πω ότι η ψηφοφορία για την έκθεση Μωράν Σαρτιέ και Ιουγγέρου έγινε με πλήρη διαφάνεια και σεβόμενη το άρθρο 59 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο προβλέπει ότι η προσωρινή συμφωνία για το ε, ποια ψηφοφορία θα προηγείται ε, ψηφίζεται σε μία ψηφοφορία εκτός και αν το Κοινοβούλιο κατόπιν ετήματος ε, μίας πολιτικής ομάδος ή ε, ε, αριθμός βουλευτών που ισούται με το 5% αποφασίσει να προχωρήσει την ψηφοφορία για τις υπόλοιπες ε, σχετικές τροπολογίες βάσει της παραγράφου 4. Το αίτημα της ομάδος ΙΕΝΕΦ να ψηφιστούν οι υπόλοιπες τροπολογίες ψηφίστηκε, απορρίφθηκε και επομένως ο πρόεδρος ε, ε, έθεσε προς ψήφιση την προσωρινή συμφωνία